The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur. We have a couple of shadows available, so so we can start. Good morning, everyone. Uh, day two of. Έχουμε τον εισηγητή, τους έχουμε όλους. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετά φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα μας επισκεφθούν και δύο υπουργοί. Έχουμε ψηφοφορίες. και αρκετά νομοθετικά κείμενα. Ξεκινάμε με την ε, πρόταση τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Συμφωνήσαμε στην προηγούμενη θητεία για αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν και δημοσιονομικές επιπτώσεις και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η τροποποίηση. Έχουμε τον εισηγητή και θα του δώσω το λόγο. Δίνω το λόγο στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ε, από τις πλημμύρες στην Ισπανία ε, και την Ιταλία μέχρι τις πυρκαγιές σε Αμαζόνιο και στην Αυστραλία την τελευταία φορά, βλέπουμε καθημερινά τις συνέπειες της, κλιμα... της κλιματικής αλλαγής. Ο νέος μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το RESC-EU που δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου έχει ως στόχο να συνδράμει τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των φυσικών και άλλων καταστροφών γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα ώστε να περιοριστούν και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, φυσικό πλούτο και ιδιωτικές περιουσίες. Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2019, επιπλέον της εθελοντικής δεξαμενής εθνικών μέσων, δημιουργήσαμε το RescueU, μια πανευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων, όπως πυροσβεστικά αεροπλάνα, ελικόπτερα και ειδικό ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Τα μέσα αυτά θα αγοραστούν από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα χρηματοδοτήσει το 80 με 90% των συνολικών εξόδων αγοράς και συντήρησης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει και το 100% των εξόδων. Θωρακίζουμε έτσι την Ευρώπη από φυσικές καταστροφέ όσο και από ιατρικά επίγοντα περιστατικά, όπω είναι μια επιδημία ή άλλου ειδών απειλών όπως είναι χημικές, βιολογικές ή πυρηνικές. Στόχος της παρούσας έκθεσης, για την οποία έχω την τιμή να παρουσιάσω σήμερα, είναι καταρχήν να διασφαλίσουμε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 21-27 ο μηχανισμός θα έχει τα καλύτερα χρηματοδοτικά εφόδια ώστε να μπορούν να γίνει η αγορά των απαραίτητων μέσων και να μπορεί να λειτουργήσει και αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό, σαν Κοινοβούλιο, πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής για ένα ισχυρό προϋπολογισμό που θα είναι τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, είναι η ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την προηγούμενη περίοδο. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία τη έκθεσή μου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτηση που είχε γίνει πριν τα Χριστούγεννα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολογούσε υπέρ της πρότασής της για διαγραφή του παραρτήματος, βάσει του οποίου μια ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού για δαπάνες πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Για λόγους όμως διαφάνειας, αλλά και προστασίας της θεσμικής ισορροπίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η επαναφορά του παραρτήματος. Δεν θα διαφωνήσουμε με την ύπαρξη πολιετών προγραμμάτων εργασίας, αρκεί αυτά να στηρίζονται. Κατανοώ τις πολύ διαφορετικές ανάγκες που προέκυψαν την τελευταία προϋπόθεση του μηχανισμού πριν από δύο χρόνια. Γι' αυτό το λόγο προτείνω την τροποποίηση των ποσοστών τόσο για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο και για την προηγούμενη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσό των δαπανών για την πρόληψη δεν καταβάλλεται μέσω του μηχανισμού, αλλά των περιφερειακών ταμείων καθώς και του Ταμείου για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Επίση, πρέπει να κατανοήσουμε την ανάγκη τη Επιτροπή για μεγαλύτερη ευελιξία. Γι' αυτό προτείνω η λύση να είναι μια παρέκκληση που μπορεί το ποσοστό να φτάσει στο 10% και την τροποποίηση των ποσοστών αυτών ώστε κατά κατά, ε, η πράξη κατά 100%. Με αυτές τις αλλαγές και αφού χρησιμοποιήσουμε τα ποσοστά που ήδη έχει προπολογίσει, νομίζω ότι ικανοποιούμε το κύριο αίτημά τη για ευελιξία, χωρί να δημιουργούμε κάποιο περιττό γραφειοκρατικό βάρο. Προβλέπουμε ακόμη να χρηματοδοτείται με του ίδιου κανόνε η αποστολή μέσων που ανήκουν στην εθελοντική δεξαμενή, ανεξαρτήτω αν αυτά χρησιμοποιούνται εντό ή εκτό τη Ένωση. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση και οι συνέπειέ τη είναι εμφανεί παντού. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να συνδράμει και σε τρίτε χώρε, όποτε αυτό το ζητηθεί, είτε για την αντιμετώπιση δυσμενών συνεπειών ενό τυφώνα, είτε για την καταστροφή ενός τροπικού δάσου, είτε οτιδήποτε άλλο επηρεάζει τον πλανήτη. Πιστεύω επίση ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση όλων των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των πολιτών. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το δορυφορικό σύστημα Γαλιλαίο και η δυνατότητα αποστολή μηνυμάτων έκτακτη ανάγκη όταν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή του. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μην αφήσουν αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών μέσω του Γαλιλαίου μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για την αποφυγή ή τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζώων. Τέλος, με τροπολογίες που προτίθεμαι να καταθέσω, θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει με τροπολογιε που δυνατότητα να προβεί στην αγορά τόσο των μέσων μαζί με, το, μαζί με τα κράτη-μέλη, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μην γίνονται από κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί, επιτυχάνοντας καλύτερους όρους. Επίσης, είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα της έμεσης διαχείρισης, όπως το είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε. Αναμένω μια επικοδομητική συνεργασία με τους κοιόδης συγητές, ώστε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα για το οποίο στο τέλος θα είμαστε περήφανοι όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Η θα πάρουν το λόγο. Ο κύριος Νούνιο Μέλο έχει το λόγο πρώτος. Η πρόταση αυτή έχει σημασία και έχει και δημοσιονομικές συνέπειες ε, για την περίοδο 17-27. Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί έχουν προβλεφθεί ανάμεσα στο 14 και στο 20. E Όταν βλέπουμε ποια είναι τα επίγοντα θέματα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη βλέπουμε ε, ποιες είναι οι ανάγκες, βλέπουμε τις συνέπειες ας πούμε των κλιματολογικών αλλαγών, βλέπουμε τις ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης. Αυτά τα ζήσαμε επίσης επανειλημμένα δυστυχώς ε, ε, και στις πυρκαγιές και στη δική μου χώρα που είχαν σοκάρει το σύνολο του υπόλοιπου κόσμου. Ε, θυμίστε πριν δύο χρόνια είχαν υπάρξει άνω των 50 νεκρών στην Πορτογαλία από τις πυρκαγιές και αυτό μας οδήγησε στο να αναγκαστούμε να ζητήσουμε βοήθεια από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν ε, που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν κάποια όρια στη συνεργασία ε, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, έχουμε τις πυρκαγιές των δασών, έχουμε τις πλημμύρες, έχουμε τα σεισμικά φαινόμενα που κάθε χώρα προσαρμόζει τις ικανότητές της σε συγκεκριμένα φαινόμενα. Ως εκ τούτου είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός ο οποίος να καλύπτει τις ανάγκες και τις ελλείψεις των κρατών μελών αναπερίπτωση. Συνεπώς λοιπόν η ενίσχυση δημοσιονομική του μέσου αυτού είναι απαραίτητη έτσι ώστε και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο ανταπόκρισης οι ικανότητες αντίδρασης του συγκεκριμένου μηχανισμού να βελτιωθούν. Επανειλημμένα βιώνουμε πλημμύρες στην Γαλλία, πυρκαγιές φοβερές στην Ελλάδα, ε, σεισμικά φαινόμενα στην Ιταλία. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον κύριο Ανδρουλάκη που ασχολήθηκε με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Καταθέτουμε κάποιες τροπολογίες που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες έτσι ώστε ο μηχανισμός αυτός να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο συνειδητοποιούμε πλήρως τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σαφής έλλειψη πιστώσεων και σε σχέση με το 13-13 του 2013. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας εξαρτάται επίσης και από την ταχύτητα ανταπόκρισης μετά τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, είδαμε ότι τελικά τα φαινόμενα αυτά είχαν προκαλέσει σχεδόν 100 νεκρούς. Πολλοί δυστυχώς είχαν καεί στα οχήματά τους, στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Περισσότεροι από ό,τι στην Αυστραλία, σε μια τόσο μικρή χώρα. Συνεπώς λοιπόν γνωρίζουμε ε, τα προβλήματα αλλά δεν είμαστε ικανοί να καλύψουμε τις συνέπειες. Και φοβάμαι ότι το σύστημα το οποίο διαθέτουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον διαθέταμε δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί. Βλέπουμε τα δάση των ευκαλύπτων στην Πορτογαλία, τα δάση των πεύκων στην Ελλάδα. Δυστυχώς καίγονται τα δάση αυτά με υψηλές ταχύτητες και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν ε, μέτρα πρόβλεψης για την αποτροπή αυτών των ε, φαινομένων. Ε, φυσικά όταν μιλάμε για απλή μοίρε σαν παράδειγμα πρέπει να έχουμε τα μέσα τα συγκεκριμένα σε χώρες που υποφέρουν όπως η Γαλλία. Όταν μιλάμε για σεισμούς τα μέσα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε χώρες όπου εκδηλώνονται σεισμικά φαινόμενα όπως η Ιταλία και αντίστοιχα για χώρες ε, που υποφέρουν από τις πυρκαγιές των δασών. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Νικόλα Στεφανιάτη, εκ μέρου τη ομάδα Renew Europe. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική παρουσίαση και να ζητήσω και να συγχαρώ και το προσωπικό που βοήθησε και την Επιτροπή για την πρότασή τη. Έχω πει πολλέ φορέ ότι η αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση είναι κάτι για το οποίο καμία χώρα δεν είναι αρκετά πλούσια να το κάνει μόνη τη. Ούτε η Γερμανία, ούτε χώρε μέχρι τη Βουλγαρία, Ρουμανία, κανεί δεν μπορεί μόνο του να το αντιμετωπίσει. Άρα είναι μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη πρόταση, την οποία χρειαζόμαστε γιατί θα φτάσουμε τον Ιούλιο και θα φτάσουμε στα κράτη-μέλη και πάλι θα έχουμε πυρκαγιέ ε, στα δάση και πάλι θα έχουμε εξαιρετικά ε, ακραία καιρικά φαινόμενα, διάφορε ε, στι ε, στις συνθήκε συνθήκες ε, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν από μήνε. Τώρα, συγκεκριμένα για την έκθεση αυτή, στο παράρτημα 1 δεν θα ήθελα αυτό να αποτελέσει εμπόδιο για όλε τι διαπραγματεύσει, διότι υπάρχει κάποια λογική σε αυτά που λένε και η Επιτροπή και ο εισηγητή. Η Επιτροπή θέλει μεγαλύτερη ευελιξία, δεν πρέπει να είμαστε άκαμπτοι ώστε να μην μπορούμε να δράσουμε όταν χρειαστεί. Και ο εισηγητή έχει δίκιο όταν λέει ότι για την ετοιμότητα και για την αντιμετώπιση χρειαζόμαστε πόρου εξοπλισμό έτοιμο και ε, όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, ούτω ώστε να μην προσπαθούμε τελευταία στιγμή κάθε φορά που συμβαίνει μια καταστροφή να βρούμε κάτι. Θα ήθελα να πω ότι ε, ε, δεν ε, μας έρχονται όλα τα καλά πράγματα όταν τα θέλουμε. Ίσως λοιπόν να χρειαστούν κάποιες διαπραγματεύσεις για το παράρτημα 1 για να γίνουμε λίγο πιο ευέλικτοι. Να προσθέσω επίσης και κάτι άλλο που ανέφερε και ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Θα θέλαμε περισσότερες δράσεις ε, για τις ε, απειλές CBRN, ε, χημικού, βιολογικού και ραδιολογικού πολέμου. Η νέα, ο νέος κλάδος της συνθετικής βιολογίας, όπου παράγονται οι οι οποίοι μπορούν να εξαπλωθούν στον πληθυσμό, είναι ένας κίνδυνος. Δεν μπορούμε να μην έχουμε την κατάλληλη ετοιμότητα και να μην έχουμε φάρμακα και φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό για να βοηθήσουμε τους πολίτες και αυτούς οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν τον ιό. Δεν μπορούμε να εκθέσουμε αυτούς που θα είναι οι πρώτοι που θα ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους πανδημίες. Είμαι από την ε, Ρουμανία και τα αποθέματα, η ανοσοσφαιρίνες είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό θέμα. Γι' αυτό ε, πρέπει να έχουμε κατά νου και την αποθήκευση ε, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Ο, επίσης, ο σύνδεσμος ε, κτηνιάτρων μου έστειλε ε, ένα μήνυμα που με ενημερώνει ότι στην Αυστραλία χρειάζονταν και ιατρικό εξοπλισμό και κτηνιάτρους επιτόπου και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέραμε να βοηθήσουμε εκεί που θα χρειαζόταν. Θα έπρεπε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το μήνυμα ότι είναι ικανή να βρίσκεται επιτόπου και ο λαό τη Αυστραλία να βλέπει την παρουσία μα. Κυρίε και κύριοι, η έκταση που ε, κάει και στην Αυστραλία, 10 εκατομμύρια εκτάρια, είναι ίση περίπου με την έκταση της Αυστρίας. Και σκέφτομαι το εξή. είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες δασικές πυρκαγιές, να καούν δηλαδή το καλοκαίρι δάση που θα έχουν την έκταση της Αυστρίας. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μας καταλάβει ανέτοιμους ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός. Όχι βέβαια και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε δράση το συντομότερο δυνατόν και γι' αυτό θέλουμε συνεργασία και διαπραγματεύσεις Νομίζω ότι γενικά υπάρχει συνένεση στην αίθουσα, εκτός από το θέμα του παραρτήματος ένα, αλλά νομίζω θα βρούμε την κατάλληλη ευελιξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων, Μαγκέν Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον εισηγητή μας, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα πολιτικής προστασίας ούτω ώστε να βελτιώσουμε την προετοιμασία μα, την ετοιμότητά μα και να είμαστε έτοιμοι για φυσικέ καταστροφέ. Και ένα βασικό στόχο είναι να μπορούμε να έχουμε μια δεξαμενή πόρων για να μπορούμε σε περίπτωση καταστροφή να έχουμε κοινού εμπειρογνώμονε και πόρου. Έγινε αναθεώρηση πέρυσι από το Συμβουλίο και από το Κοινοβουλίο και χαίρομαι για το μηχανισμό Rescue. εφόσον η εθελοντική δεξαμενή δεν δίνει επαρκή πόρους. Το Rescue δείχνει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία κατά των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών και των ανθρωπογενών καταστροφών κάποιες φυσικές καταστροφές είναι ανθρωπογενείς λόγω της αλλαγής του κλίματος. Θα προτιμούσαμε να έχουμε χρηματοδότηση από νέες πηγές, ωστόσο δεν συμφώνησε το Συμβούλιο σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν τώρα με αυτό το μηχανισμό ανακατανομής να τα βγάλουμε πέρα. Θεωρούμε σημαντικό ε, να έχουμε ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή, ιδίως βλέποντας τις καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειαζόμαστε αύξηση των πόρων. Επίσης, χαίρομαι διότι ο εισηγητής ε, ε, ε, μιλάει για το επόμενο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου θα πρέπει να παραμείνει το ποσό για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ε, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα επαναφοράς του παραρτήματος στο κείμενο, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό για τις ομάδες αντιμετώπισης και για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. για δραστηριότητε και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε επίσης και τη χρήση του συστήματος Γαλιλαίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία για το θέμα αυτό μαζί με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκ Ανδριώστο, εκ μέρους του e ε, ναι, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω και ξέρετε ότι έρχομαι από την Ιταλία, άρα δηλαδή για μας η, ε, πολιτική προστασία είναι καθοριστική σημασία. Μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτό το μηχανισμό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα και για κάποιε τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Και εγώ θέλω να πω ότι το παράρτημα 1 ε, πρέπει λιγάκι να το σκεφτούμε, όχι γιατί θέλω να είμαι εχθρικό, αλλά κυρίω γιατί θέλω να υπογραμμίσω αυτά που είπε κυρίω η Επιτροπή, η οποία προτίθεται να διαγράψει το παράρτημα αυτό, ε, γιατί υποτίθεται ότι θα βοηθήσει περισσότερο στο περιεχόμενο. Αλλά και εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει ε, με αυτή την κίνηση να θίξουμε κάποια βασική μας αρχή. Ε, πιστεύω ότι κάπου θα βρούμε κάποια λύση. Ε, ακόμα και η πρόταση να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικά προηγμένα συστήματα από το σύστημα Γαλλέως ε, και αυτό το συμμερίζομαι. Όπως σας είπα, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής προστασίας της Ιταλίας είναι το να δρά κανεί με ταχύτητα και αυτό οφείλεται κυρίως στην ε, περιφερειακή οργάνωση και στο συντονισμό. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε, να μιμηθούμε κάποια συστήματα που έχουν αποδειχθεί χρήση χρήσιμα στα κράτη-μέλη. Ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες. Ελπίζουμε να μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτές τις τροπολογίες, γιατί με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε ομοφωνία. Θεωρώ ότι το θέμα της ε, πολιτικής προστασίας, όπως είπαν όλοι, δηλαδή η ασφάλεια των ανθρώπων και των αντικειμένων της περιουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να επιτύχουμε δυνατόν μια ομόφωνη στάση. Για το ECR δεν βλέπω να υπάρχει σκιώδη ηγητής, που σημαίνει ότι περνάμε στην ΓΚΟΕ. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Η υπεθέρμανση του πλανήτη και συνεπώς οι κλιματολογικές αλλαγές είναι πλέον κάτι το σταθερό και δυστυχώς αυξάνεται η συχνότητα και η ένταση ε, σπάνιων στο παρελθόν φαινομένων. Είδαμε τις τρομερές πυρκαγιές ε, στην Αυστραλία, ε, επίσης είδαμε τις συνέπειες με τις καταιγίδε άμμου στην ίδια χώρα, προβλήματα επίσης στην Ινδονησία. Υπάρχει μια αλληλουχία καιρικών φαινομένων που δημιουργούν προβλήματα. Συνεπώς λοιπόν ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να γίνει κατανοητός σαν μια απαραίτητη προσπάθεια προσαρμογής στα νέα φαινόμενα. Και ο εισηγητή πολύ σωστά επιμένει σχετικά με την ανάγκη 1,4 δις για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση της διασυνοριακής ανταπόκρισης και συντονισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τα μέσα στις νέες ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το Rescue ε, μέσω της χρήσης άλλων ε, δυνατοτήτων που έχουμε όπως τον Γαλιλαίο και εδώ είναι η ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση κυρίως με την εξωτερική διάσταση των φαινομένων αυτών. Ευχαριστώ τον εισηγητή, θα στηρίξουμε την πρότασή του και ελπίζω να υπάρξει σε αυτό το σημαντικό θέμα ομοφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουν οι εισηγητές. Τώρα περνώ στα μέλη της Επιτροπής. Stuart David. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα είμαι σύντομη, έχετε πάρα πολλά θέματα μπροστά σας, λέει η πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να, πω από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή πόσο σωστά είναι τα νέα στοιχεία τα οποία προτείνει ο εισηγητή, ιδιαίτερα σχετικά και με το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση του Καλλιλέου όπως επίσης και την δυνατότητα ε, χρηματοδότησης επιχειρήσεων εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των μέσων αυτών. Το είδαμε πέρυσι για τη Μοζαμβίκη και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης είδαμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι κανόνες ε, του μηχανισμού αυτού σε σχέση με την ταχεία αντίδραση να είναι απλή. Θα ήθελα να ελθώ κυρίως στο παράρτημα υπαρίθμου 1. Δεν είναι γραφειοκρατικό το θέμα, είναι λειτουργικό. Αντικειμενικά έχει σαν στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις διατάξεις για το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ και να ενισχύσει την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοια φαινόμενα. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές επενδύσεις σε τομείς όπως καταπολέμηση των πυρκαγιών ή της παροχής υψηλού επίπεδου εξειδίκευσης ιατρικών υπηρεσιών, εκένωσης περιοχών και ε, άλλα θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Θα πρέπει λοιπόν να, να διασφαλίσουμε μάλλον ότι ο προϋπολογισμός που θα καλύψει τις επενδύσεις αυτές ε, περιέχεται στις διατάξεις που ήδη υπάρχουν στο παράρτημα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μέγιστη δυνατή ευελιξία ε, πάντα κρατώντας την ισορροπία της διοργανικής συμφωνίας να υπογραμμίσω το ότι πράγματι ελπίζουμε η φιλόδοξη πρόταση για 1,4 δις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο να υποστηριχθεί και να στηρίξει τις προσπάθειες για την πολιτική προστασία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το συνολικό ποσό το οποίο θα είναι διαθέσιμο για την πρόληψη και ανταπόκριση, η απόκριση, θα αυξηθεί φυσικά και αυτό. Συνεπώς λοιπόν σε αυτά τα ποσοστά που προτείνεται θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να επενδύσουμε από κοινού στις ικανότητες αυτές και στα μέσα αυτά και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων έτσι ώστε να κάνουμε επιτέλους το επόμενο βήμα σε επίπεδο πολιτικής προστασίας εμείς λοιπόν θέλω να καταθέσουμε εκκλήσεις για περαιτέρω ε, αυξημένη ευελιξία και υποστηρίζουμε την ουσία της πρότασης ε, που περιέχεται στο παράρτημα 1. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις μέσω τροπολογιών που αφορούν το δημοσιονομικό κομμάτι και οι οποίες διασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή ευελιξία και την κοινή προμήθεια εξοπλισμών. έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε με σωστό τρόπο τις πιστώσεις οι οποίες ε, θα τεθούν στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια συνένεση και για το παράρτημα η συζήτηση δεν έχει κλείσει. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Για τις απόψεις που κατέθεσαν ε, για το ζήτημα του Rescue είναι όλες χρήσιμες και είναι σημαντικό ότι οι περισσότεροι από εμά, για να μην πω όλοι, προερχόμαστε από χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ζητούν οι πολίτες των χωρών μας, τι ζητούν οι πολίτες Ευρώπης και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να πετύχουμε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα οδηγήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του Rescue, ώστε ένας μηχανισμός λειτουργικός που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις της επόμενης περίοδου. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες, ώστε μετά να ανοίξει αυτή η συζήτηση με ένα γόνιμο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And indeed, as the rapporteur has said, the deadline for amendments... Ευχαριστώ πολύ. Ε, προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών 28 Ιανουαρίου και στις 5 Μαρτίου προβλέπεται για την ε, απόφαση στην Επιτροπή και αργότερα ελπίζω το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειο Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος ε, είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό, ο οποίος φτάνει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Καλημέρα Πασκάλ. Άρχισα να λέω αυτά τα οποία θα έλεγες εσύ και έφτασε στην κατάλληλη στιγμή για να σου δώσω το λόγο. Okay, thank you uh, again for to Tobias for opening the meeting and sharing the opening of the meeting. Uh, ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ ο συμπρόεδρος ουσιαστικά. Θα θέσουμε το θέμα του Brexit λοιπόν. Όπως γνωρίζετε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή θα στείλει τη δική της γνωμοδότηση στις αρμόδιες επί της ουσίας, ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με ένα νέο τρόπο πλέον στο Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε το θέμα όχι μόνο σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά το πώς από εδώ και πέρα να δούμε τι έχει γίνει και σε σχέση με τη διαπραγμάτευση μέχρι σήμερα. Η επιστολή αυτή είναι μια τυπική μεν διαδικασία, αλλά είναι και η έναρξη, θα έλεγα, της πολιτικής συζήτησης για το τι θέλουμε να περιλαμβάνονται, να περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις ε, για τα εμπορικά θέματα. Ο Λίζε από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το λύπηρο. Πολλοί από εμά ε, θα στεναχωρηθούμε ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει ή μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς η συμφωνία αυτή είναι καλύτερη από το να υπήρχε έξοδος ε, χωρίς συμφωνία στο τέλος του μήνα. Είναι ένα πρωτοθετικό θέμα ε, να ξέρετε ανοργάνωτο Brexit θα είχε πάρα πολλά θέματα, συνέπειες, προβλήματα, ελλείψεις σε φάρμακα κτλ. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια συμφωνία, αλλά η συμφωνία ε, φυσικά απλά μας οδηγεί στο τέλος του χρόνου αυτού και αν δεν μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά ε, το πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί σε περίπτωση μη συμφωνίας μπορεί να αναφανεί εκ νέου στο μέλλον. Και η μακροπρόθεσμη συμφωνία, η εμπορική με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι το οποίο ε, ε, είναι απαραίτητο και έτσι και αλλιώς το τέλος του χρόνου δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε όλα πολλά θα μείνουν σε εκκρεμότητα, τα ιατρικά υλικά και εξοπλισμοί, η κατάσταση των ασθενών. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να συνεργαστούμε και σε θέματα ε, κλιματολογικά. Εδώ έχουμε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επόμενη κόπ γίνεται στη Γλασκόβη. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να πετύχει και εμείς επίσης. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες, να έχουμε ένα κοινό όραμα στην κλιματολογική πολιτική. Και ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ε, καθιστούμε απόλυτα σαφές ότι θα θέλαμε τα θέματα του περιβάλλοντος και του κλίματος ε, να βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια διάταξη και τώρα και κατά την επόμενη χρονιά, όπως ακριβώς ανέφερε ο Πίτερ. Εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών ε, θεωρούμε ότι είναι ανησυχητικό το να διαπιστώνουμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο και από την άλλη πολιτικές ε, δηλώσεις. Τα θέματα του κλίματος μπαίνουν στις πολιτικές δηλώσεις και αυτό αποδυναμώνει το περιβάλλον ε, τουλάχιστον κατά τα επόμενα ετή και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι όταν ε, ε, συζητάμε για το τι είναι σημαντικό για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, εμείς ως σοσιαλδημοκράτες αυτό το θέμα το βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ μεγάλη χώρα μεγάλος πληθυσμός, βρίσκονται δίπλα μας, ε, συνεργαστήκαμε για τόσα πολλά χρόνια και τώρα ενδεχομένως να αναγκαστούμε να ακολουθήσουμε διαφορετική ε, κατεύθυνση για θέματα περιβάλλοντος. Και εάν συμβεί αυτό, Ας μην ε, ξεχνάμε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία αγορά δίπλα μας ε, που θα έχει λιγότερες ε, προσδοκίες για το περιβάλλον, για θέματα κλίματος, προστασίας από την κλιματική αλλαγή. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται δίπλα μας Βεβαίως ε, μπορούμε ε, να ασκήσουμε πίεση στα Ηνωμένα Έθνη, στη Βραζιλία, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάμε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δίπλα μας, είναι γείτονά μας και ό,τι κάνει θα επηρεάσει τη δική μας την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε λοιπόν να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτά όλα που σας λέω περιλαμβάνονται στην πολιτική δήλωση. Δεν φτάνει αυτό και αυτά που διαβάζουμε και αυτά είναι απλά ε, ευχολόγια. Ε, δεν είναι μια συμφωνία που να επιβάλλει υψηλέ προδιαγραφές για το κλίμα και για το περιβάλλον. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στην όλη συζήτηση. Από κοινού να διασφαλίσουμε ότι αυτά που υπάρχουν δεν αρκούν, ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλότερε φιλοδοξίες για το κλίμα και το περιβάλλον. Και θα ήθελα βεβαίως να επισημάνω και προς όφελος των πολιτών και όσων εξαρτώνται από τα φάρμακα ότι πρέπει να επισημάνουμε και το θέμα της αλυσίδας εφοδιασμού για φάρμακα για να μην προκύψει μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν σημαντικά φάρμακα για την υγεία τους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν έχω να πω πάρα πολλά μετά τον Πίτερ και τη Γιούτα. Νομίζω ότι ε, όλους μας ενοχλεί λιγάκι η διαδικασία κατά το μάλλον ήτον το βρετανικό πολιτικό σύστημα μοιάζει να έχει ε, χάσει τον έλεγχο όπως ε, φαίνεται και οι πυρκαγιές ε, στην Αυστραλία. Υποτίθεται έχουμε τώρα μια συμφωνία αλλά το θέμα είναι ε, πού θα είμαστε μετά από 11 μήνες. Ε, όσοι προσεύχεστε το βράδυ, μην ξεχνάτε να περιλαμβάνετε στην προσευχή σας ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να βοηθήσουμε τους Βρετανούς ε, να βρουνε μια διέξοδο. Κατά κάποιον τρόπο το οικολογικό θέμα στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι τόσο κακό όσο σε άλλα κρατημέλη, γιατί οι Βρετανοί δεν χρησιμοποιούν πια τόσο πολύ τον άνθρακα. Αυτό είναι η καλή πλευρά ε, της υπόθεσης. Από την άλλη βέβαια έχουμε περιοχές, μεγάλες περιοχές, όπου έχουμε βιομηχανία που δεν λειτουργεί πια, ένα οικονομικό σύστημα ε, με πολλές ε, ανομαλίες και όλα αυτά ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ε, πολιτικές ε, περιπέτειες, περίπου όπως τα έχουμε ήδη διαπιστώσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να σώσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μπάς και τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο αίσθημα συμμεριζόμαστε για το Brexit και με κάποιους βρετανου συναδέλφους, όχι σε όλες τις πολιτικές ομάδε, αλλά σε ορισμένες πολιτικές ομάδε. Γνωρίζοντα ότι η συμφωνία αποχώρηση θα εγκριθεί μάλλον από το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και το Brexit θα γίνει στι 31 Ιανουαρίου, τώρα αρχίζει η πραγματική δουλειά γιατί μιλάμε για τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολλά θέματα που είναι πολύ σημαντικά και βρίσκονται στο πεδίο αντικειμένου της Επιτροπής μας για όλους τους σχετικούς κανονισμούς, φάρμακα, ιατρικές συσκευές, όλα αυτά έχουν κέρια σημασία για τις μελλοντικέ μας σχέσεις και μας απασχολούν και μας ανησυχούν. Στι διαπραγματεύσει αυτέ θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι στι μελλοντικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο Ιδίω για το περιβάλλον, θα πρέπει να ακολουθεί τη σχετική νομοθεσία. Δεν θέλουμε να έχουμε μια Σιγκαπούρη στον Τάμεση δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει όλους να μας ανησυχεί και αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Πολλοί λένε ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Το πολιτικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο αν σπρώχνει προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των συνομιλίων σε ένα χρόνο, ανησυχώ πάρα πολύ για ένα άτακτο Brexit. Η γνωμοδότηση την οποία θα δώσουμε ως Επιτροπή ΕΝΒΗ πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και η πραγματική δουλειά ξεκινάει μετά τη Συμφωνία Αποχώρησης γιατί τότε θα διαμορφώσουμε τις μελλοντικές μας σχέσεις στις οποίες θα πρέπει να φροντίσουμε πάρα πολύ την τήρηση της νομοθεσίας μας, την πρόσβαση σε φάρμακα κλπ. Άρα τώρα ξεκινάει η δουλειά. Εκ μέρους των ID, θέλετε εσείς το λόγο, δεν έχουμε κάποιο ομιλητή. Κύριε Μάκιντάρ, για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα αποτελέσματα του Brexit είναι ότι τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία που έχω να μιλήσω στην Επιτροπή και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Το κείμενο που έχουμε τώρα είναι ισορροπημένο και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και χαίρομαι που έχουμε αυτό το καλό κείμενο. Θα προσπαθήσω να ε, απαλύνω κάποιους από τους φόβους σχετικά με την απομάκρυνση από τους κανονισμούς, ιδίως σε ε, σχέση με τις δράσεις για το κλίμα και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπος στις παραγράφους 5 και 6. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας από τους ε, πρωτοπόρους στη δράση για το κλίμα και μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από τις ρυθμιστικές πρακτικές και της χώρας μου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα εμπορία εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η πρώτη ε, παγκόσμια εφαρμογή αυτού του συστήματος ξεκινήσαμε το 2002, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την εφαρμογή του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η χώρα που ε, προσπαθούσε τα τελευταία δέκα χρόνια να ζητήσει ε, μεταρρυθμίσεις για να έχουμε μια σωστή τιμολόγηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να βοηθήσει το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάλαμε την τιμολόγηση των ε, ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για να βοηθήσουμε. Και τον ε, Ιούνιο του 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη μεγάλη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο που υιοθέτησε νομοθεσία για να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 και είναι πολύ γερά τα θεμέλια. Οι εκπομπές στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώνονται σταθερά από ε, το νόμο του 2008 ε, για την ε, αλλαγή του κλίματος. 44% χαμηλότερες από το επίπεδο του, 2000, του 1990 ήταν οι εκπομπές, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακου στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο χρόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και πολύτιμο εταίρος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να διδαχθούμε αμοιβαία και να βάλουμε τις οικονομίες μας στο σωστό μονοπάτι για την απαλλαγή από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Βλέποντας λοιπόν το μέλλον, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα επικεντρωθεί σε πολιτικές με βάση επιστημονικά δεδομένα, κάτι το οποίο τα τελευταία οκτώ χρόνια έχω προσπαθήσει, έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε όσο είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω ότι οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάζουν πολύ πιο προσεκτικά και πολύ πιο θετικά θέματα όπως ε, γονιδιακή τεχνολογία και οι γενετικά, και τους γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Και ίσως ε, οι Γάλλοι γεωργοί θα μπορούν να αγοράζουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς τους από την άλλη μεριά της μάχης και όχι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το Brexit πράγματι είναι ε, κάτι το ιδιαίτερα λυπηρό, αλλά είναι πλέον ένα δεδομένο. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες στον τομέα των φαρμάκων, στον τομέα των ρυθμίσεων για το περιβάλλον και επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα γύρω από την συνέχιση της ε, επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση στις διαπραγματεύσεις και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να χαλαρώσουν οι περιβαλλοντικές συμφωνίες οι μελλοντικέ συμφωνίες στον τομέα του ελευθέρου εμπορίου θα επηρεάσουν ιδιαίτερα ε, την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ελπίζω η συμφωνία να είναι μακρόχρονη, να βοηθήσει στην σταθεροποίηση ε, της προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς η συμφωνία Μερκοσούρη είναι το παράδειγμα προς αποφυγήν εδώ Ελπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορέσει να συνεργαστεί στις ε, συμφωνίες ε, τις οποίες ε, έχουμε μπροστά μας. Η ΚΟΠ στη Γλασκόβη είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να αποτύχει, έχει σημασία και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρει δυνατότητες σε μας και ως Επιτροπή και ως θα έλεγα πολιτικοί άνδρες και γυναίκες να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις συμφωνίες τις περιβαλλοντικές που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τις μορφές διαλόγου πλέον με τους συναδέλφους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα δώσω το λόγο σε δύο συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ λέει η κυρία Φίλιπς που μου δίνετε το λόγο που είναι και η τελευταία φορά. Ελπίζω κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο να επανέλθει. Αυτά τα θέματα θα έλεγα είναι σημαντικά όχι μόνο για την Ένωση αλλά και για, την, για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσο Βρετανίδα Ευρωβουλευτής ανησυχώ για, τις, ε, για τους προσανατολισμούς του ε, Μπόρις Τζόνσον που ε, διαφοροποιεί την πορεία της χώρας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται θα χρησιμοποιήσουν την συμφωνία απόσυρσης έτσι ώστε να μειώσουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι αναφορές στη Συμφωνία των Παρισίων και στην αρχή ε, του όποιος μολύνει πληρώνει έχουν αφαιρεθεί από το πρωτόκολλο συμφωνίας. Είναι κρίσιμο το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ε, σε επίπεδο συμφωνίας ε, στο εσωτερικό των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία αυτή η οποία έρχεται οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι για να αποφύγουμε μια κατάρρευση του κλίματος δεν έχουμε πάνω από δύο, δέκα χρόνια μάλλον μπροστά μας. Ήδη ε, χτες ε, η συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας ε, συμφώνησε με την Σκοτία και την Ουαλία εναντίον των ρυθμίσεων που προτείνει η κυβέρνηση του Λονδίνου τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου λοιπόν διαφωνούν και δεν δίδουν την πολιτική εντολή στην κυβέρνηση του Λονδίνου για να κάνει πραγματικότητα τις προτάσεις της. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάντα η δυνατότητα μη συμφωνίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Γνωρίζουμε από το κρυφό έγγραφο που κυκλοφόρησε τι σημαίνει αυτό έλλειψη στα φάρμακα, αύξηση των τιμών, μείωση της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών. Είναι μια ανόητη η διαδικασία αυτή και έτσι οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από τη Βρετανία είναι καταδικαστές. Η Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επιστολή που είναι ισορροπημένη και θίγει τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εγώ συμμερίζομαι αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι ότι είναι μια επικίνδυνη συμφωνία και ακολουθούμε έναν επικίνδυνο δρόμο και μακάρι να μην είχαν γίνει όλα αυτά όπως και οι άλλοι συνάδελφοι από το ECR Υπάρχει το θέμα της ε, ανταλλαγής εκπομπών, αλλά Θέλω να σας πω ότι ανησυχώ λιγάκι. Η συντηρητική κυβέρνηση έχει δείξει με σαφήνεια ότι το περιβάλλον για αυτήν δεν είναι προτεραιότητα. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα όσο θα θέλαμε. Ε, μιλάμε για τη γραφειοκρατία και ε, πώς ε, το Brexit ε, δίνει τη δυνατότητα ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύσει όλη αυτή την ε, ενωσιακή νομολογία και κανόνες και να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Αυτό εμένα με ανησυχεί, γιατί φοβάμαι ότι το πρώτο που θα κάνουν είναι να ξεφύγουν από αυτό που εκείνοι αποκαλούν γραφειοκρατία. Εμείς όμως λέμε ότι είναι πρότυπα ασφαλείας, παραδείγματος χάρη για τα τρόφιμα. Και είδαμε στα, στο θέμα των συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν τα πρότυπα και στις δύο πλευρές. Για μένα το θέμα της ασφάλειας τροφίμων με ενισχύει πάρα πολύ. Ε, κοτόπουλα με χλωρίνη, το έχουμε δει το πρόβλημα. Επίσης, μιλήσαμε για ακαδημαϊκές έρευνες. Νομίζω αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Μαζικά φεύγουν οι ακαδημαϊκοί από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Και τι θα γίνει τελικά με τους ακαδημαϊκούς. Ε, και νομίζω η φήμη μας ε, σε αυτό το χώρο θα χάσει πάρα πολύ ριζικά. Το θέμα των ιατρικών μηχανημάτων τα παρεμφερεί, ε, εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν τελικά να διαπραγματευτούν για αυτό το θέμα και δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με την πρόσβαση σε φάρμακα στον Ρωμανό Βασίλειο. Πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Ελπίζω η Επιτροπή Περιβάλλοντος να μπορέσει να ασκήσει επιρροή σε οποιαδήποτε συμφωνία τελικά επιτευχθεί. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω τελειώνοντας, λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριος Πάλμερ. Και εγώ προφανώς ε, συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που ελέγχθησαν από τους ε, συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις ε, πολιτικές ομάδες. Εγώ ένα θέμα θέλω να προσθέσω. Είναι μάλλον η τελευταία φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και θέλω να πω ότι όσες δυσκολίες και αν προκύψουν απογοήτευση για το Brexit και όπως και οι συνάδελφοί μου και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το δρόμο που αρχίζει να ακολουθεί η χώρα μου. Εν πάση όλα όσα μπορεί και αν παρουσιαστούν λόγω της συμφωνίας αποχώρησης, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι στην Επιτροπή Υγείας, ε, γενικότερα σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα έρευνας, που είναι αποφασισμένοι κάθετα αποφασισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσουν τη στενότερη δυνατή σχέση με τους συνεργάτες και φίλες μας εδώ. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ίσως να φεύγουμε από τις επίσημες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, η επιθυμία να παραμείνουμε κοντά, να συνεργαστούμε, αυτή η επιθυμία δεν έχει χαθεί και δεν θα χαθεί. Εγώ οποτεδήποτε θα συναντώ έρευνες που ασχολούνται παραδείγματος χάρη για θέματα καρκίνου για μακροχρόνιε ε, ασθένειε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι θέλουν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με του εταίρου του ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε τελειώντα, θέλω να πω ότι για μένα ήταν ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφου, τη Γραμματεία και του συμβούλου τη δική μου τη πολιτική ομάδα. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ε, καλή τύχη, σας εύχομαι τα καλύτερα στις μελλοντικές σας προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έλεγα επισήμως να τους χειροκρατήσουμε όλους τους Βρετανούς συναδέλφους μας. Thank you. We... Ευχαριστώ. Δύο λεπτά σύντομο διάλειμμα πριν τις ψηφοφορίες.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 για την ε, λεγόμενη ταξονομία σε εισαγωγικά. Υπήρξε μια πολιτική συμφωνία το Δεκέμβριο, αλλά θα πρέπει να επικυρωθεί επίσημα με τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ. Στις 9 την Πέμπτη λοιπόν. Μην το ξεχάσετε. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία. Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ηλεκτρονική ψήφος. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Συνεπώς η επιστολή της Επιτροπής μας ε, γίνεται δεκτή και θα αποσταλεί. το αντίρρηση σχετικά με την παρουσία μολύβδου στο PVC. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η αντίρρηση γίνεται δεκτή και θα επανέλθει το θέμα στην Ολομέλεια. Δεκατέσσερα. Τροπολογία 50. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 63 υπέρ, κατά, δεκτή. 65 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 67 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 66 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές τα περίφθη 70 υπέρ κατά υπέρ πάλι κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τοπολογία 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 85 υπέρ κατά έλεγχος 85 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές δε, απερίφθη. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 90 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 91 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 92 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 93 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 94 υπέρ, κατά, αποχές απε... δεκτή. 96 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές δεκτό 99 υπέρ κατά αποχές δεκτό 100 υπέρ κατά αποχές δεκτό 101 υπέρ κατά αποχές δεκτό 102 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 103 υπέρ κατά αποχές δεκτό 104 υπέρ κατά αποχές δεκτό 105 υπέρ κατά αποχές δεκτό 106 υπέρ κατά αποχές δεκτό 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 και 3 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6. 7 μάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 9 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 10 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 12 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 13 ή μάλλον 14 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18 υπέρ. Συγγνώμη, το 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας προφορίες. Δεκτή. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική τελική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συγχαρητήρια στη διαπραγματευτική ομάδα. Και περνάμε στην ψηφοφορία για το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης, του 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Πράσινων Πόλεων. Τροπολογία 54, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνω, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την 56. Πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. μαζί με την 63 ψηφίστηκε. Ε, Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80-84 αποσύρονται, 85 ψηφίζουμε υπέρ, Κατά. Ας το ελέγξουμε για την 85. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 85. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε για την 87. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. Για την 92. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, 95. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε για την τροπολογία 9. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά. Ας το ελέγξουμε για τη 16. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε και πάλι για την 18. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και την 20. Εγκρίνεται. Αν δεν σας πειράζει, ας κάνουμε και τη 19 που δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 19. Την προηγούμενη, γιατί δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 19. Και περνάμε στην 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τη 45. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε τη 47. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τη 49. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 50. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο, για το σύνολο του ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Συγχαρητήρια λοιπόν.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το σύνολο της απαλλαγής άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η απαλλαγή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο στις ψηφοφορίες για τις ελάχιστες απαιτήσει ε, για επαναχρησιμοποίηση του νερού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίνεται η θέση την οποία ακολουθήσαμε στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, περιμένοντας τον Υπουργό της Κροατίας σε περίπου 15 λεπτά.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, πολλά θέματα, πολλές ερωτήσεις για σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια παρουσίασή σας δεκάλεπτη, μπορείτε να εκθέσετε τις προτεραιότητές σας και μετά θα ακολουθήσουν δύο γύροι ερωτήσεων. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Προσδοκώ μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Το επόμενο εξάμεινο θα ηγηθεί η χώρα μου των προσπαθειών για τη Συμφωνία των Κρατών Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα του περιβάλλοντος με κάθε αμοιβαίο σεβασμό. Βρισκόμαστε σε μια εποχή διεθνούς αβεβαιότητας, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και ελπίζουμε η μεταβατική περίοδος να γίνει πραγματικότητα με επιτυχία. Έτσι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και την ενότητα που πρέπει να μας χαρακτηρίζει στους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει προωθώντας κοινέ αξίες και κοινέ πρωτοβουλίε για όλα τα κράτη-μέλη. Μια ισχυρή Ευρώπη στον τομέα του περιβάλλοντος ε, μας οδηγεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες. Αναπτυσσόμενη Ευρώπη, διασυνδεδεμένη Ευρώπη, Ευρώπη που προστατεύει και ισχυρή Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Στην αναπτυσσόμενη Ευρώπη θέλουμε μια ουδέτερη κλιματολογικά ανάπτυξη, βασική προτεραιότητα της κρατικής Προεδρίας, είναι το Ευρωπαϊκό Green Deal, η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα το 50 και προσαρμογή στις συνέπειες ε, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες, ε, βρισκόμαστε λίγο πριν ε, το σημείο, θα έλεγα, ανεπανόρθωτης βλάβης. Απαιτείται λοιπόν κατεπίγουσα δράση. Αναγνωρίζοντας την κρίση αυτή, ελπίζω να κρατήσουμε υψηλά τους στόχους που έχουμε. Η στρατηγική ατζέντα για το 2019 μέχρι το 2024 και το Ευρωπαϊκό Green Deal στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου, σύμφωνα και με τους στόχους της COP Παρισίων, καθορίζει, θα έλεγα, την πορεία μας για τα επόμενα χρόνια. Η Κροατική Προεδρία θα ξεκινήσει το Συμβούλιο της Εργασίας για τη Green Deal και όπως προτείνεται και στην αρχική σας αντίδραση την προηγούμενη εβδομάδα Συμμεριζόμεθα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Green Deal είναι μια νέα στρατηγική ανάπτυξη μετατρέποντας την Ευρώπη σε μια ευημερούσα και ισχυρή οικονομικά κοινωνία και σε μια ανταγωνιστική οικονομικά κοινωνία στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των πόρων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και προστασίας και έλογης χρήσης των φυσικών πόρων. Ε, το να πετύχουμε τους στόχους του Green Deal απαιτεί ε, επενδύσεις και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνουμε εμείς ε, το πρόγραμμα δράσης για την αηφόρο Ευρώπη που παρουσίασε η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ θέσεις σε νέους τρόπους χρηματοδότησης, έτσι ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή κλιματολογική ουδετερότητα. Να διευκολύνουμε την μετάβαση σε μια αποδοτική σε επίπεδο κόστους και ωφέλιμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας θα κάνουμε συζητήσεις για το Green Deal σε όλες τις συζητήσεις και στο ΕΚΟΦΗΝ τον Ιανουάριο ε, και τον Φεβρουάριο ε, και το Συμβούλιο για την Νεότητα και τον Ιούνιο ε, και για τα θέματα πολιτισμού κτλ. Ελπίζουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε συζητήσεις και για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις τις οποίες θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις αυτές θα δείξουν τους τομείς τους οποίους απαιτείται να υπάρξουν αλλαγές στην βιοπικιλότητα στην προστασία, στους τρόπους προστασίας της βιοπικιλότητας. Θα υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές και δεν θα υπάρξουν απαράδεκτοι συμψηφισμοί. Τώρα, η, κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Κροατίας θα δούμε ακριβώς τι μπορεί να κάνει η ε, Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η αηφόρος οικονομία. Τώρα για τις δραστηριότητες μας στα πλαίσια της μετρίασης ε, των συνεπειών των αλλαγών του κλίμα, θα προωθήσουμε στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και να προωθήσουμε επίσης για τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της μείωσης των εκπομπών. Αυτά εγγράφονται στα πλαίσια της πολιτικής μας σε σχέση με τις εκπομπές ε, για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να υποβάλουμε τις νέες μας προτάσεις στην αρμόδια, στο αρμόδιο πάνελ των Ηνωμένων Εθνών το ταχύτερο, δυνατότητα, ταχύτερο δυνατό. Ταυτόχρονα η βιοπικιλότητα είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε. Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη βιοπικιλότητα μετά το 2030 έτσι ώστε να Διοθετήσουμε μετά από το 2030 ένα νέο πλαίσιο βιοποικιλότητας και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα δημοσιευθεί το Μάρτιο είναι καλοδεχούμενη. Και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας που ζητάει μια φιλόδοξη πολιτική και φιλόδοξους στόχους και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχοι της Προεδρίας είναι να υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για να διευκολύνει την πρόοδο των θεμάτων αυτών και στην Ένωση και στα διεθνή φόρα και να συνεχίσουμε και την προετοιμασία για το COP15 στην Κίνα. Να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη είναι αφιερωμένα στην προσπάθεια διατήρησης της ηγέτιδας θέσης της Ένωσης σε σχέση με ένα ρεαλιστικό αλλά και φιλόδοξο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προκαλέσει τις απαιτούμενες αλλαγές άμεσα και έμεσα αντιμετώπισης της απώλειας βιοπικιλότητας και την προώθηση της βιοπικιλότητας σε όλους τους οικονομικούς τομείς, όπως και στα πλαίσια της ΚΟΠ των Παρισίων. Η Ένωση θα πρέπει να είναι ηγέτιδα στις δράσεις της. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα συνεχίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύει και να στηρίζει τις προσπάθειές μας στον τομέα των βιοποικιλότητας. Τώρα σχετικά με την τελευταία προτεραιότητές μας, σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα φαινόμενα μόλυνσης στα πλαίσια της νέας μετάβασης. Ε, θα πρέπει με τη νέα διαχείριση των αποβλήτων να προχωρήσουμε επίσης σε αλλαγές και σε σχέση με τις συσκευασίες και ε, διάφορα μέτρα πρόληψης της θαλάσσιας μόλυνσης. Να μου επιτρέψετε επίσης ε, να προχωρήσουμε και να σας αναφέρω τα νομοθετικά βήματα τα οποία σκοπεύουμε να κάνουμε για αυτά τα οποία είναι σε ε, κρεμότητα. Πρώτον, ε, η κατάληξη των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό. Όταν γίνει αυτό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, με το Κοινοβούλιο. Για τα MRV ε, επίσης οι συζητήσεις συνεχίζονται για τα νέα θέματα. Θα ξεκινήσουμε συζητήσεις ε, για τις πρώτες νομικές ρυθμίσεις, ε, νομικές επαναλαμβάνω ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κλίματος και των κλιματολογικών αλλαγών λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπάρχοντα προγράμματα και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος λήγουν στο τέλος του 2020. Περιμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα ανάμεσα στις, στα δύο προγράμματα. Για τα μη νομοθετικά θέματα θα δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια του Green Deal για την κυκλική οικονομία είναι μια απαραίτητη τροποποίηση θα έλεγα της οικονομίας μας στα πλαίσια α, της οικονομικής μας ανάπτυξης. Ε, το Συμβούλιο θέλει να υιοθετήσει συγκεκριμένα συμπεράσματα στον τομέα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και ε, στα πλαίσια της επανεξέτασης των νομοθετικών υποχρεώσεων που υπάρχουν και των σχετικών νέων προτάσεων μέσα από το Green Deal θα οργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων σε υπουργικό επίπεδο για τους ελέγχους που γίνονται και την αξιολόγηση της διαχείρισης ε, των υδάτων σε ε, όλες τους τις μορφές. Αγαπητά μέλη, θα κλείσω λέγοντας ότι η Κροατική Προεδρία θα είναι αφιερωμένη πλήρως και θα προωθήσει όλα τα θέματα τα οποία προανέφερα στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Green Deal. Θα προωθήσουμε λοιπόν τις ε, φιλοδοξίες τις οποίες έχουμε εκφράσει για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοπικιλότητας και την χειροτέρευση του περιβάλλοντος είναι κοινό στόχος, είναι κοινή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για, την, για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι επίσης μια νέα ευκαιρία για μια ευημερούσα, αναπτυσσόμενη και πετυχημένη Ευρώπη. Προσδοκώ σε σωστή συνεργασία μαζί σας, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Να περάσουμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ένα συμμετέχον από κάθε πολιτική ομάδα. Από το ΕΛΚ καταρχήν, ο Πέτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ένα βασικό θέμα. Η Προεδρία σας ε, θα πρέπει να ασχοληθεί με το βασικό αυτό θέμα της ε, προστασίας ε, του κλίματος για να επιτύχουμε τους στόχους για το 2050 και το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές συμφώνησε το Δεκέμβριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το στόχο, η δική μας πολιτική ομάδα τουλάχιστον. στο Συμβούλιο είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να σας ζητήσω τη δική σας εικόνα για το στόχο για το 2030. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευρία η υποστήριξη. Η πλειοψηφία λέει ότι ε, θα πρέπει να φτάσουμε στο 55% χωρίς προϋποθέσεις. Ε, η δική μας ομάδα υποστηρίζει τη στάση της Επιτροπής, μιλάμε για το 50% και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το 55% να φτάσουμε και πιο πέρα. Δεν ξέρω αν στο Συμβούλιο υπάρχει πλειοψηφία για το 50% καν. Γι' αυτό θα θέλαμε τη δική σας πολιτική εικόνα. Πώς βλέπετε την κατάσταση, πόσο έχουμε προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και για μας στο ΕΛΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμά του το ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις διεθνείς πτυχές και θα ήταν θαυμάσιο αν όλοι οι συμβαλόμενοι και οι Ηνωμένε και η Βραζιλία, όπου έχουμε και άλλες δυσκολίες, αν όλοι εξέφραζαν τις φιλοδοξίες τους ε, κατά 10% υψηλότερα σε σχέση με τη Συμφωνία του, του Παρισιού. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να καταβάλλετε προσπάθειες και γι' αυτό. Και αφού αναφέρατε και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, για μα είναι πολύ σημαντική η έρευνα. 120 δισεκατομμύρια ευρώ για την ουδετερότητα του κλίματο, για βιομηχανία που να είναι ουδέτερη ω προ το κλίμα. Αυτό προωθεί και η δική μα πολιτική ομάδα. Είστε έτοιμοι να προωθήσετε αυτού του στόχου ε, που προωθεί και το Κοινοβούλιο για να επιτύχουμε την ουδετερότητα για το κλίμα και με βάση τι τεχνολογικέ εξελίξει Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Λουένο. Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε? Δύο λεπτά, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε. Είναι σημαντικά τα θέματα που αναφέρατε, όχι μόνο η κλιματική αλλαγή που είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε και όλα τα υπόλοιπα. Παραδείγματος χάρη την νομοθεσία που απαιτείται για την παράνομη ξυλία και τα προϊόντα της και το κατά πόσο θα μπορούν να απολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, άλλη μια ερώτηση τι προτίθεται να κάνει η δική σας Προεδρία για το θέμα της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ούτως ώστε να πληρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές και η οδηγία πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων. Είναι φιλόδοξη η πρότασή σας για την αναθεώρηση αυτών των ε, οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την, ε, τις αεροπορικές μεταφορές, νομίζω ότι θα συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εκπομπή αερίων άλλων εκτός του διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης, ε, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου θα πρέπει να κλείσουμε το θέμα της έγκρισης τύπου για τα εμπορικά οχήματα και τα ελαφρά οχήματα και να ασχοληθούμε και με τον προϋπολογισμό, γιατί χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. και η Επιτροπή Περιβάλλοντος πολλές φορές συζητά την ε, περιβαλλοντική φορολογία θεωρητικά περισσότερο παρά πρακτικά. Δεν ξέρω αν η Προεδρία σας έχει κάποια ξεκάθαρα θέματα, κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τη φορολογήση για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ομάδας Ρήνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Με εντυπωσιάζουν ορισμένοι από τους στόχους της Κροατίας. Ιδίως για την ε, ομάδα ποδοσφαίρου και την ομάδα μπάσκετ που έχετε σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν όμως ε, μιλάμε για τους περιβαλλοντικούς σας στόχους για τους επόμενους έξι μήνες, δεν εντυπωσιάζομαι εξίσου με τις αθλητικές σας επιδόσεις, γιατί αν δείτε την νομοθεσία για το κλίμα, παραδείγματος χάρη, για να επιτυχούμε κάτι πριν από τη διάσκεψη κορυφής με την Κίνα, πριν από το COP26, κάτι θα πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει να φα ε, σαν center for στο, στο ποδόσφαιρο και να μην είστε απλώς αμυντικός παίκτη. Θα ήθελα λοιπόν να ενισχύσετε την προσέγγισή σας. Είπατε ότι θα διεξαχθούν συζητήσεις. Καλές είναι οι συζητήσεις. Αλλά αυτό που θα ήθελα να δω εγώ είναι το Συμβούλιο να παίζει ρόλο center force σε τέτοια θέματα. Μπορεί να μην σας αρέσει η δική μου προσέγγιση, αλλά εμείς οι Βόρειοι είμαστε πολύ ξεκάθαροι με τις θέσεις μας για τέτοια προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις πολύ φιλόδοξες απαντήσεις σας για να σηκώσω και εγώ την κροατική σημαία και να σας υπερασπίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόλγκρεμ εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και για τις φιλόδοξες ε, παρουσιάσεις σας. Ω επιστήμον για θέματα που έχουν σχέση με το κλίμα, ελπίζω ειλικρινά ότι θα προωθήσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα ώστε να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις απαιτήσεις των επιστημόνων για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Έχουμε ακούσει τις συζήτηση για το 50-55% αλλά τα επιστημονικά δεδομένα μας δείχνουν 70% ότι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε ε, ε, να κάνουμε κάτι και θα πρέπει να αρχίσουμε ήδη από φέτο και από του χρόνου να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Μια ερώτηση συγκεκριμένα τώρα για την Κροατική Προεδρία. Ε, επειδή ξέρω ότι έχετε ως χορηγό μία πετρελαϊκή εταιρεία, την IAM, και ε, ε, σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις αυτό δημιουργεί ζήτημα. Δεδομένου του ρόλου της Προεδρίας υπάρχει ένας κίνδυνος, η χορηγία να θεωρηθεί ότι επιτρέπει επιρροή σε αυτή την εταιρεία επί της ευρωπαϊκής ε, θέσπισης νομοθεσίας. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτή τη δήλωση η οποία πλήττει το γόητρο της Κροατικής Προεδρίας. Πιστεύετε ότι δεν πειράζει να έχετε ως χορηγό μια πετρελαϊκή εταιρεία για την Προεδρία σας όταν ε, επικεντρώνεστε στην Πράσινη Συμφωνία και στην εξάλληψη των ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρίζιν, εκ μέρους του IND. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως αναφέρετε πολύ σωστά στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η μαζική, και η μαζική μείωση της βιοπικιλότητας είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές αυτοκαταστροφικά, μερικές φορές από ιδεαλισμό προσπαθεί ε, να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με τη Συμφωνία του Παρισιού θα βάλουμε ένα στόχο ουδετερότητας έναντι του άνθρακα που δημιουργείται εξή ζητήματα. Ποιο θα είναι το μερίδιο των πυρηνικών ε, ε, σταθμών της πυρηνικής ενέργειας Ποιε θα είναι οι κυρώσει που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση ε, αθέτησης των υποχρεώσεων των κρατών. Θα υπάρχουν παρεκκλήσει στο σύστημα αυτό. Και τέλος, οι στόχοι αυτοί πώς συνδυάζονται με την επιβίωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που είναι ζωτική σημασία για την οικονομία μας. Η επιτυχία, κύριε Υπουργέ, θα εξαρτηθεί από την κυριαρχία και τη διατήρηση της κυριαρχίας των κρατών μας και τη διατήρηση της κυριαρχίας στο έδαφος τους, αντί να έχουμε μία γραφειοκρατία που θα μας ισοπεδώνει όλους. Θα πρέπει πολύ συχνά να το υπενθυμίζουμε αυτό, γιατί τα κράτη θα πρέπει να έχουν την κυριαρχία επί των νόμων τους και την γνώση επί του εδάφους τους, γιατί μόνο έτσι μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά. Ξέρουμε ότι όλες αυτές οι καταστροφές που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να δράσουμε. Για το ECR, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, εμεί είμαστε συντηρητικοί ε, και στηρίζουμε ανεπιφύλακτα όλα αυτά που γίνονται για το περιβάλλον, ε, για το καθαρό αέρα, την καθαρή ατμόσφαιρα, προστασία της βιοπικιλότητας. Βέβαια, έχουμε κάποιες ε, αμφιβολίες και επιφυλάξεις ε, όσον αφορά την κλιματική πολιτική. Υπάρχουν ε, δύο επιφυλάξεις. Το ένα αφορά στην ταχύτητα με την οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία. Δηλαδή, η πρόταση είναι να εγκριθεί ε, ο νόμος περί κλίματος το καλοκαίρι ε, φέτος ε, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και παρά το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αξιολόγηση για να προχωρήσουμε στους στόχους του 2030 και αυτή η αξιολόγηση δεν θα έτοιμη πριν από το καλοκαίρι. Τέλος υπάρχει και ένα νομικής φύσεως ε, θέμα ε, κατά πόσον ε, μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν υπάρχει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο. Και το άλλο θέμα αφορά στα κονδύλια που χρειάζονται για να διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την επένδυση 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ε, παραμένει ένα πολύ μεγάλο ποσό και ως εκ τούτου όλα εξαρτώνται και από τα αποτελέσματα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάρα πολλά εξαρτώνται και από τους ιδιώτες επενδυτές. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω η Προεδρία πώς ακριβώς τοποθετείτε απέναντι σε αυτήν την κριτική που ε, λέει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές παραχωρήσεις και παρόλα αυτά δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο μακροχρόνιος ε, προϋπολογισμός. Και τελευταίος ομιλητής, πριν σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Υπουργέ, η Κροατική Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια πολύ προβληματική περίοδο και τα ερωτήματα που καλείστε να απαντήσετε είναι καθοριστικής ε, σημασίας και για το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουμε να τα καταφέρετε. Υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να θίξω παρότι βλέπω ότι είστε αρκετά φιλόδοξοι στην ημερήσια διάταξή σα. Πρόκειται για την ε, κλιματική ουδετερότητα και για την ε, προστασία της ε, βιοπικιλότητας. Και θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο πώς ακριβώ αποφασίζει για την ουδετερότητα σε σχέση με τις πλαστικές ύλε. Μέχρι το 2050 κατ' ουσίαν προβλέπεται ομοφωνία μόνο για τα μεμονωμένα μέτρα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική απόψη. Η ουδετερότητα ε, σχετικά με τους υδρογονάνθρακες είναι σημαντική και η στρατηγική πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ε, μέχρι το 2030 αρκούν αυτά που γνωρίζουμε επιστημονικά το 50% δεν αρκεί, αλλά ούτε και το 55%. Υπάρχουν ε, επιστημονικά δεδομένα και έχουμε και την αρχή της ε, πρόληψης. Το ε, λιγότερο θα έπρεπε να έχουμε 60% για να έχουμε κάποια ασφάλεια. Αν λοιπόν μέχρι το 2030 δεν υπάρχουν επαρκείς δεσμεύσεις, ε, νομίζω ε, θα πρέπει μετά να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι και αυτό ε, θα είναι πολύ δαπανηρό. Ποια είναι τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας για να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να καταλήξουμε όσον αφορά στην βιοπικιλότητα. Ελπίζω να έχετε μια στρατηγική η οποία θα είναι μια πραγματική αντίδραση σε αυτή την έκτακτη κατάσταση. Η ε, προστασία της, ε, των ειδών ε, είναι καθοριστική σημασία για την επιβίωση στον πλανήτη μας. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στην αυξανόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Πολύ ωραία. Ε, είσαστε έτοιμος για να απαντήσετε. Έχετε 10 λεπτά. Poštovane dame i gospodo, hvala Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα που θέσατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα με τη σειρά που ετέθησαν. Ε, κάποια ερωτήματα βασικά είναι παρεμφερή. Ε, ως εκ τούτου θα τα συνενώσω διάφορα ερωτήματα. Υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι αναφέρθηκαν ε, στο θέμα της, ε, του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής, αλλά καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν ετέθη το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο για μια συμφωνία 55% μέχρι το 2030. Αν δεν απατώμε, το ερώτημα αυτό ετέθη από τον κύριο Λίζε. Και ε, την ίδια κατεύθυνση ακολούθησε και το τελευταίο ερώτημα που ετέθη από την κυρία Μούντικ προς την ίδια λοιπόν κατεύθυνση. Γνωρίζετε ότι αυτό θα το ε, καταλάβουμε τον Ιούνιο εάν τελικά και όταν μάλλον θα γίνει ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Οι στόχοι της ε, Κροατικής Προεδρίας είναι μετά την παρουσίαση της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και αυτό ελπίζουμε να γίνει το Μάρτιο, να ξεκινήσει μια συζήτηση ε, σε όλα τα επίπεδα και κατόπιν τον Ιούνιο να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια στον δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο. Οι Υπουργοί ε, Περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να υπάρξει αγώνας για την κλιματική αλλαγή. Και όλοι γνωρίζουν επίσης ότι σε αυτόν τον αγώνα ε, κατά της κλιματικής αλλαγής δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση. Ως εκ τούτου και η δική μας η απόφαση για την ε, κλιματική αλλαγή, ε, η δική μας η απόφαση για την Πράσινη Συμφωνία και αυτή δεν έχει εναλλακτική, αυτή είναι η μόνη λύση. Και ελπίζω αυτό να φανεί κατά τους επόμενους μήνες και στις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Κατόπιν, ε, κυρία Μούντικ, ίσως μπορώ να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Εσείς ε, διερωτηθήκατε πώς μπορεί κανείς να επιβάλλει στα κράτη-μέλη να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Ίσως θα πρέπει τώρα όμως να κάνω μία γενικότερη τοποθέτηση για να απαντήσω αυτό το ερώτημα, να μιλήσω γενικότερα για την Πράσινη Συμφωνία. Αυτό το έγγραφο ε, αποδεικνύει ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Και αυτό ισχύει και για όλους τους άλλους που ακολουθούν το δικό μας το παράδειγμα. Έτσι λοιπόν αυτό θεωρώ ότι είναι και ο μόνος σωστός δρόμος τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε, δηλαδή ε, μια υποχρέωση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να μπορούμε να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να εξηγήσουμε στα κρατη ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τίποτα για τις υποχρώσεις τους. Ε, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι αυτά τα κάνουμε για μας τους ίδιους και για τις μελλοντικέ γενιές. Εδώ λοιπόν λοιπόν θέλω ε, να τοποθετηθώ και σε αυτά που είπε ο κύριος Τόμπαλτς και σε αυτές τις αλληγορίες που ανέφερε σχετικά με τον αθλητισμό. Κύριε Τόρβαλτς, ε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς οι Κροάτες ε, δεν μιλάμε πολύ για τον αθλητισμό, κάνουμε περισσότερο πράγματα στον αθλητισμό. Ως εκ τούτου, όσον αφορά την δική μας την δέσμευση σε σχέση με την κλιματική νομοθεσία, να είσαστε σίγουροι ότι και εκεί θα κάνουμε πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο επιθυμώ να μεταφέρω με κάθε σαφήνεια και ελπίζω και το μήνυμα αυτό να το εισπράξετε εσείς ως ε, Ευρωβουλευτές. κατόπιν στο θέμα της ε, τεχνολογικής ε, πρόοδου ή των ε, προσπαθειών που είναι απαραίτητες έτσι ώστε αυτή η τεχνολογική πρόοδος να πετύχει και να μπορούμε να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι πρικοδοτημένη με κονδύλια και αυτό που ενδιαφέρει είναι να βρούμε απλώς τις ε, απαραίτητες ε, πλατφόρμες. Και για την τεχνολογική πρόοδο εμείς προτείνουμε νέες δυνατότητες, ε, όλα αυτά ελπίζω να συμπεριληφθούν στο πολιτευστημο δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίως στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι απαρέγκλητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε την τεχνολογική πρόοδο και ως εκ τούτου και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Όσον αφορά στο μέλλον της Ευρώπης και γενικότερα στο μέλλον του κόσμου, ε, αν δούμε το θέμα του κλίματος, εκεί τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί κανείς ε, να εξετάζει τις διάφορες χώρες αποκομμένα. Και βεβαίως εμείς ε, εξετάζουμε το θέμα της ε, κυριαρχίας ε, κάθε χώρας, εθνικής κυριαρχίας, αλλά όταν πρόκειται για το κλίμα, το περιβάλλον, το μέλλον μας, νομίζω εκεί πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη ως ένα σύνολο και να ε, δρούμε όλοι από κοινού. Ίσως αυτό να έχει στα αυτιά σας αφελές, αλλά ειδικά τώρα, τώρα που βρισκόμαστε όλοι εδώ και συζητάμε, υπάρχουν διάφορα ε, κλιματικά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη στην Κροατία έχουμε την ε, χειρότερη ατμόσφαιρα των τελευταίων ετών. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι κάνει κρύο και χρησιμοποιούμε τη θέρμανση. Τι να πω τώρα στους ε, Κροάτες, ότι ξέρετε αυτά είναι το από αποτέλεσμα ε, ενεργειών πολιτών από άλλες χώρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο κλίμα επηρεάζει μία χώρα την άλλη. Βεβαίως ε, και διαφυλάσσεται η εθνική κυριαρχία, αλλά συγγνώμη, όταν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, η εθνική κυριαρχία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, εκεί η Ευρώπη πρέπει να δρά από κοινού. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει ε, να καταλήξουμε σε συνένεση για τα βασικά θέματα τα οποία επιθυμούμε να προάγουμε και να προωθήσουμε ε, τους επόμενους έξι μήνες. Όσον αφορά στην οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας ή αν θέλετε την ερώτηση του κ. Λουένου, Βεβαίω και έχει μεγάλη σημασία να έχουμε καλή ποιότητα ατμόσφαιρας, ε, υδάτων ε, και ε, οικοσυστήματα που να συνδέονται μεταξύ τους. Στη συνεδρίαση του Μαρτίου θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων αναλύσεις και αξιολογήσεις των υδάτινων πόρων και εκεί θα ληφθούν και αποφάσεις σε σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας, με βάση όλα αυτά που προείπα, γνωρίζετε ότι αυτή η συζήτηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Υπουργών Περιβάλλοντος, αλλά κυρίως στις αρμοδιότητες των Υπουργών Οικονομικών, όπου γίνονται διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο. Και κατόπιν υπάρχει και το θέμα του ότι μερικές χώρες ε, ε, εναντιώνονται στους ε, στόχους της πράσινης ε, συμφωνίας. Συμφωνία υπάρχει ε, για τους στόχους του 2030. Ε, κατά τα άλλα, όλα τα άλλα πρέπει να επιληθούν σε ανώτερο επίπεδο. Εμείς στο δικό μας το Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να υπάρξει μία περαιτέρω συζήτηση, να υπάρξει ως δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία, να ε, να προσπαθήσουμε για την ε, κλιματική αλλαγή και για την Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί ως ε, ηγέτιδα δύναμη σε αυτόν τον αγώνα για την κλιματική αλλαγή. Ετέθη επιτάπητος και το θέμα των εναέριων μεταφορών. Ε, υπήρξε μια συγκεκριμένη ερώτηση από αυτού. Αυτή τη στιγμή οι εκπομπές από τις εναέριες μεταφορές αντιστοιχούν στο περίπου 3% του συνόλου των εκπομπών και θεωρούμε ότι οι εναέριες μεταφορές θα πρέπει και αυτές να εξεταστούν για να μειωθούν οι εκπομπές μέχρι το 2050. Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο, αλλά βέβαια μην ξεχνάτε ότι και πάλι εδώ εμπλέκονται θέματα φορολογικά, εισφορών, άρα δηλαδή πάει και αυτό το θέμα στις αρμοδιότητες των Υπουργών Οικονομικών. Κατόπιν ετέθη το θέμα της ε, διατήρησης των ειδών και βιοπικιλότητας. Εμείς ε, επ' αυτού θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σημαντικό έγγραφο. Γνωρίζουμε ότι η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα πρέπει να δημοσιευτεί τους επόμενους ε, έξι μήνες και ε, όταν θα έχει δημοσιευτεί αυτή η στρατηγική τότε και εμείς θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε να αναπτυχθούν επιχειρήματα σε αυτή τη στρατηγική. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο αγώνας για την διαφύλαξη της ε, βιοπικιλότητας ε, συνδέεται άμεσα με τον αγώνα για την κλιματική αλλαγή, άρα ε, και τα δύο θέματα απαιτούν την προσοχή μας, όπως επίσης και η νομοθεσία για το κλίμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά σε σχέση με το χρονισμό, θα θέλατε εσείς να υπάρξει μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο τον Ιούνιο. Καλά, δεν είναι, δεν είναι υποχρέωση αυτό που θα αναλάβετε, αλλά είναι ο στόχος σας. Στρατηγική μας και στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να προχωρήσουμε μέχρι τον Ιούνιο για το νομικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτός είναι ο, η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. Περιμένω και άλλες ιδέες γύρω από αυτό. Καθώς περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων, με το ΕΛΚ πάλι. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Ήταν ενδιαφέρουσα η εισαγωγή την οποία κάνατε. Υπάρχει βέβαια το θέμα της χρηματοδότησης του Green Deal. Ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η πρόθεσή σας έτσι ώστε να πετύχουμε ένα κάποιος, μια κάποια συνένεση. Υπάρχουν εδώ εμπλεκόμενοι φυσικά και οι Υπουργοί ε, Οικονομικών. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια ικανοποιητική μέθοδο χρηματοδότησης του Green Deal. για τη σοσιαλιστική ομάδα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Άκουσα τις φιλοδοξίες σας και την βούληση την οποία εκφράσατε έτσι ώστε να διευκολύνετε την προσπάθεια για το νομική ρύθμιση για το κλίμα και άκουσα αυτό που είπατε ότι θα κάνετε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε και να μην μείνουμε μόνο στα λόγια. Το εκτιμούμε αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εδώ, το οποίο πολλοί συνάδελφοι στην Επιτροπή αυτή έχουν ήδη θίξει ίσως. Είναι η ατζέντα την οποία έχετε μπροστά σας για φέτος. Έχουμε την COP στη Γλασκόβη, έχουμε την COP15 στην Κίνα για τη βιοπικιλότητα, έχουμε τη συνάντηση κορυφής Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωση το δεύτερο εξάμεινο. Συνεπώς λοιπόν η Προεδρία σας καθίσταται κρίσιμη για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συναντήσεων, για τη διαχείριση σωστά αυτών των συναντήσεων. Οι παρασκευαστικές συναντήσεις θα γίνουν το πρώτο εξάμεινο, το τρέχον εξάμεινο, και τουλάχιστον για την ΚΟΠ Γλασκόβης θα πρέπει να καθαρίσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο θέλουμε. Ξέρουμε ότι για τα MBC απαιτείται μεγαλύτερη φιλοδοξία από τα κράτη-μέλη αν θέλουμε να τηρήσουμε τις συμφωνίες των Παρισίων και γνωρίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη εκπεφρασμένη επιθυμία προόδου ε, μετά από τη συνάντηση της Μαδρίτης. Είδαμε ότι υπήρχαν από πλευράς μας πολλοί δισταγμοί, σχεδόν εμπόδια. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς σκοπεύετε να προετοιμάσουμε για την συνάντηση κορυφής με τους Κινέζους έτσι ώστε να διατηρήσει την ηγετική της θέση η Ένωση στη Γλασκόβη και να δείξει ε, τις υψηλές φιλοδοξίες που έχουμε για τα MBC. σε επίπεδο ε, της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω ότι οι ερωτήσεις σας δεν πρέπει να ξεπερνούν το ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο για την Προεδρία σας, μια Προεδρία με μεγάλα θέματα και μεγάλες προκλήσεις. Ε, πρέπει να μείνω στο λεπτό. Θα θέσω δύο ερωτήσεις πολύ συνοπτικά για τον κλάδο της βιοπικιλότητας. Την προηγούμενη εβδομάδα υιοθετήσαμε ένα φιλόδοξο ψήφισμα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούμε να υπολογίζουμε με την υποστήριξη της Κροατικής Προεδρίας, έτσι ώστε η επόμενη στρατηγική βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει 10% αύξηση του προϋπολογισμού, ειδικά για την προστασία της βιοπικιλότητας, γιατί το 20 έχει ε, προβλέψει μόνο το 8,6, ε, θα έλεγα το πιο χαμηλό ποσοστό από το 14. Είναι δύσκολο να μιλάμε για μεγάλες φιλοδοξίες ε, με μικρούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς λοιπόν, οι ελλείψεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη οδηγεί στην απώλεια εκατομμυρίων ευρώ θα ήθελα να μάθω αν έχετε μία στρατηγική για τη βελτίωση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, Ευχαριστώ για το ΕΛΚ. Ο κύριος Βυσίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Υπάρχουν ε, ε, πολλοί στόχοι. You might know the EU access uh, to Danube Convention and to Elpan. Και υπάρχουν ε, πάρα πολλά διαμάντια στο περιβάλλον και πολλά από αυτά και σε περιοχές όπως τα Καρπάθια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα πρέπει ε, να ληφθούν για να έχουμε καλύτερη συνεργασία για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην περιοχή των Καρπαθίων, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. επίση, θα βελτιώσουμε την εικόνα των περιοχών ε, αυτών που είναι ιδιαίτερη εικόνα. Η ερώτησή μου είναι αν νομίζετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα εξετάσει η Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάντελ Μόζα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Περισσότερο θα μας χαροποιούσε αν ήταν λίγο περισσότερο λεπτομερές και ακριβές το πρόγραμμα και μας μιλούσατε για το ε, αν η προεδρία σας είναι κοντά στο στόχο του 50-55%. Θα υπάρξει ένα σχέδιο δράση ε, για την κυκλική οικονομία το Μάρτιο. Θα υποβληθεί από την Προεδρία σα. Μπορείτε να μα πείτε τι αναμένετε από αυτό, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό στην Επιτροπή μα ιδίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Πρασίνων, κυρία Πάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μα. Έχουμε μόνο ένα λεπτό. Θα είμαι σύντομη το ψήφισμα για την COP15 που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα προβλέπεται το 10% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας, πω, να σας ρωτήσω αν χαιρετίζετε αυτό το ψήφισμα και αν υποστηρίζετε το ότι πρέπει πραγματικά να δώσουμε χρήματα και όχι να μιλάμε απλώς και να έχουμε ε, απλά λόγια. Ε, εφόσον δεν τηρούνται οι στόχοι της βιοποικιλότητας, ε, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε τους λόγους. Δεν ε, αποκαταστάθηκαν οι κίνδυνοι και δεν τηρήθηκαν αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει. δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για τους στόχους της βιοπικιλότητας και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε αν θα υποστηρίξετε την Επιτροπή ούτως ώστε η νέα προσπάθεια για τη βιοπικιλότητα να μπορέσει να ορθοποδήσει. Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον που εκδόθηκε το Δεκέμβριο αναφέρεται η προοπτική για το 2020 και υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τη βιοπικιλότητα. Θα ήθελα όλοι να διαβάσουν την έκθεση αυτή. Υπάρχει και στο διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ζώνη που περνάει και από την Κροατία δεν προστατεύονται όλες οι περιοχές σε αυτή την πράσινη ζώνη. Θα προσπαθήσετε το έργο αυτό να γίνει ένα εμβληματικό έργο για να μπορεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχυρίζεται ότι έχει ηγετική θέση για τη βιοπικιλότητα. Εκ μέρους του ID, η κυρία Μπένιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πριν από έξι μήνες ε, ήμασταν πάλι εδώ και συζητούσαμε με τον Υπουργό της Φινλανδίας. Κάναμε την παραδοσιακή ανταλλαγή απόψεων όπως σε κάθε αρχή νέας Προεδρίας από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να ζητάμε κάποιο απολογισμό μετά από έξι μήνα και δεν θέλω να ασκήσω κριτική κατά της Φινλανδίας. Ξέρω ότι οι προεδρίες με την εξάμεινη ανάλλαγη είναι περισσότερο συμβολικές παρά πολιτικής σημασίας. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές σας για το επόμενο εξάμεινο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολλά, ε, αλλά πολύ συχνά ε, λόγω των ε, ομάδων πίεσεων, των ομάδων πίεσης, δεν γίνονται αρκετά όπως θα έπρεπε να γίνει για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπως επίσης και για την για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, ποια θα είναι η θέση της Κροατικής Προεδρίας για τα θέματα αυτά και τι προτίθεται να κάνει για να γίνει κάποια πρόοδος επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, κυρία Μπέντελε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, σας ε, συγχαίρω καταρχήν ε, που αναλάβατε την Προεδρία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Έκλεισε το μικρόφωνο. Δυστυχώς έκλεισε το μικρόφωνο η μιλήτρια. Λυπάμαι. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus dem Kommissionsvorschlag oder vielleicht auch θα με ενδιέφερε ε, ποια είναι τα θέματα εκείνα που τα βρίσκετε καλά ως κορατία, ποια είναι δύσκολα για σας ε, ε, και εσείς προσωπικά τι θα προσθέτατε σε αυτό. Και ο πρόεδρος, μικρόφωνο παρακαλούμε, με κλειστό. Εντάξει, τώρα ακούμε. Λοιπόν, το δικό μου το ερώτημα είναι το εξής. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε καλύτερα για την Κροατία, για αυτή τη χώρα. Και το ερώτημά μου είναι, ε, κατά την άποψη της ε, Κροατίας, ε, ποια είναι τα σημεία εκείνα που την ενδιαφέρουν στην πρόταση του Κοινοβουλίου της Κομισιόν για την Πράσινη Συμφωνία. Και εσείς προσωπικά, τι θα προσθέτατε σε όλα αυτά ως Κροατία. για το ECR, παρακαλώ. Κυρία Ζαλεύσκα, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, ξέρετε να δίνετε γενικές ε, απαντήσεις, γιατί είστε πολύ καλοί διπλωμάτες, αλλά εγώ ε, θα κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Κατά τους επόμενους έξι μήνες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ε, περίοδο που πρέπει να προετοιμάσουμε κάθε εβδομάδα ξεχωριστά. Θα έχουμε πολλές συναντήσεις στην Κροατία, Υπουργικά Συμβούλια και πολλά άλλα. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το πότε θα λάβουν χώρα όλες όλες αυτές οι συναντήσεις και επίσης ε, να μας πείτε κατά πόσον ε, θα πράξουν οι για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλάμε για περισσότερα χρήματα, περισσότερους φόρους. Θα ήθελα να γνωρίζω τις πληροφορίες από εσά τον ίδιο. Εσείς είσαστε ο Υπουργός ε, Περιβάλλοντος Ενέργειας και έχετε σπουδάσει οικονομικά. Ε, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει εσείς για όλες αυτές τις συναντήσεις κατά τους επόμενους έξι μήνες. Για το Renew παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα ε, στα σλοβενικά. Ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας. Η Πράσινη Συμφωνία και οι συνέπειε του είναι βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κροατία έχει συμπεριλάβει και τα Δυτικά Βαλκάνια στις προτεραιότητες. Με ενδιαφέρει πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις προτεραιότητες πώς να συνδυάσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια και το περιβάλλον. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ρήπανση στις χώρες αυτές, χώρες ε, που είναι και φτωχές. Ένα, ε, ένας παράγων ε, μεγάλης ρήπανσης είναι τα έξι οι 6 σταθμοί ενέργειας, οι 16 συγγνώμη, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ε, που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα άνθρακα. Πώς ε, θα προχωρήσει η κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην πολιτική της έναντι των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί χωρίς καθαρή ατμόσφαιρα σε αυτή την περιοχή δεν θα είναι καθαρή ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αφορά και τη γειτονική, τις γειτονικές χώρες, τη δική σας χώρα και εμάς, τη Σλοβενία. Ελπίζω ότι η Κροατική Προεδρία θα αντιμετωπίσει και αυτά τα προβλήματα σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκρατές, κύριε Ρανάη. Ο κύριο Ρανάη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Όσον αφορά την ουδετερότητα του κλίματος, θα πρέπει να δούμε τα πολιτικά στοιχεία και ε, θα πρέπει να δούμε ότι αυτό κοστίζει και πολλά χρήματα. Χωρίς ε, ισχυρή βούληση δεν θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Δέκα χρόνια μετά την αρχή της οικονομικής κρίσης, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε δώσει υψηλή αξία στο θέμα της Πράσινης Συμφωνίας, ούτως ώστε να είναι μια δίκαιη συμφωνία. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Τι εγγύησει μπορείτε να προτείνετε ούτως ώστε να μην πληρώσουν το τίμημα οι φτωχότεροι. Επίσης, άλλη μια ερώτηση ποιες είναι οι εγγυήσει που θα μπορούσαν να δώσουν τα κράτη-μέλη ούτω, ώστε τα θέματα αυτά να έχουν κοινή αντιμετώπιση και να μην προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε μεμονωμένα συμφέροντα. Θα πρέπει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφεληθεί από αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. E, Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον ε, Υπουργό κύριο Τσόλτης για την παρουσίασή του. Και εγώ έχω μια παρόμοια ερώτηση. Η Προεδρία σας ε, είναι η πρώτη Προεδρία στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας. Επίσης, ε, ε, θα οργανώσετε και μια διάσκεψη κορυφή για τα Δυτικά Βαλκάνια και αναφέρθηκε και προηγουμένω ε, η ρήπανση στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν 16 ε, σταθμοί που ρηπαίνουν και που κλείουν περισσότερο διοξίδιο του θείου από ότι όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα θέμα στη διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων και θα έπρεπε να αρχίσουμε να το συζητάμε στα πλαίσια του μηχανισμού της δίκαιης μετάβαση και μια δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας ε, για την, ε, το να συμπεριλάβουμε ε, τους στόχους SDG, ιδίως το στόχο 7 και 15. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίσιτς για τους μη γραμμένους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι το 2050 η ατριετική θα έχει καταλήξει ένας υπόνομος. Και για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά και λόγω της μεγάλης ποσότητας των πλαστικών που προέρχονται κυρίως από ε, καταναλωτικά προϊόντα στον τομέα των τροφίμων το 50% της μόλυνσης των θαλασσίων ε, αυτών περιοχών ε, προέρχεται αποκλειστικά από τις υπηρετικές περιοχές. Συνεπώς λοιπόν τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, εσείς στη χώρα σας τι σκοπεύετε να κάνετε γύρω με τα θέματα αυτά. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δυστυχώς είναι πεπαλαιωμένα. δεν επαρκούν τα μέτρα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και λόγω της διαφθοράς η οποία δυστυχώς κρατεί και στη δική σας χώρα και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας έχετε αναλάβει την υποχρέωση ε, συνολικά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσετε τη χρηματοδότηση των πολιτικών αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών και να διευκολύνετε τα μεταβατικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία αν λάβουμε υπόψη μας ότι για κάθε επενδυόμενο ευρώ σε επίπεδο πολιτικών μέτρων εξοικονομούμε 6 ευρώ τα οποία θα πρέπει εκ των υστέρων να πληρωθούν. Ακούσαμε πολλές προτάσεις γύρω από όλα αυτά. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που είπε ο συνάδελφος για το Μούρα Ντράβα στην Κροατία. Έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στην Κροατία και θα πρέπει η Προεδρία και η κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει την κατάσταση. Ο συνάδελφος Τόρβαλντ είπε ότι η Κροατία είναι καλή στον αθλητισμό. Στο κλίμα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει σαν εθνική ομάδα θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα παίξει επίθεση και ποιος κέντρο, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι ότι θα πετύχουμε. Πώς θα οργανώσετε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο γύρω από το EGB, λέει η ομιλήτρια. Thank you. So we can discuss ε, sports with you, Croatian Minister. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τον αθλητισμό, αλλά δεν μπορείτε ε, να αλλάξετε το αποτέλεσμα ε, του τελικού του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Κροατία. Έχετε το λόγο. Okay. Bilo je jako Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τουλάχιστον όσο μπορώ περισσότερες. Ε, κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένες ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση του Green Deal, σαν παράδειγμα τέθηκε από πολλούς ομιλητές. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το επιπλέον 10% για τη βιοπικιλότητα. Το έθεσε και η κυρία Ροντρίγκε και άλλοι βουλευτές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος δεν μπορεί να επηρεάσει την τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το ε, δημοσιονομικό. Αυτό όμω το οποίο μπορούμε να κάνουμε και ελπίζω να το πετύχουμε είναι να βοηθήσουμε σε εθνικό επίπεδο να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη χρηματοδότησης του προγράμματος που περιλαμβάνεται στο Green Deal. Γι' αυτό λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα έρθω σε επαφή μου και με τους ομολόγους μου σε επίπεδο Υπουργών Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να πιέσουν και τους Υπουργούς Οικονομικών και να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι σημαντικό. Το θέμα της μετρίασης και του ελέγχου των κλιματολογικών συνεπειών είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί από όλου ότι έχει πρωτεύουσα σημασία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως ένας ενιαίος τομέας τόσο σημαντικός όσο αυτός. Αυτή είναι η αντίληψη η οποία θα μας χαρακτηρίζει ε, καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας και όχι μόνο την αρχή. ήρθα εδώ ε, σήμερα και δεν μπορώ να σας δώσω εγγυήσει φυσικά ότι θα βρεθούν όλες οι απαιτούμενε πιστώσεις. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους υπουργούς περιβάλλοντος, για να κατανοήσουν οι υπουργοί των άλλων τομέων πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό σχετικά με το περιβάλλον. Και γι' αυτό ακριβώς απαιτούνται περισσότεροι δημοσιονομικοί πόροι. Τέθηκαν επίσης ερωτήσεις για τη θέση μας σε σχέση με τον Green Deal, τη θέση της κρατικής κυβέρνησης. Να σας πω ότι δεν έχει σημασία το τι πιστεύει πραγματικά η Κροατία. Εμείς προεδρεύουμε του Συμβουλίου στην παρούσα φάση και όπως γνωρίζετε ε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών. Πάντως η Κροατία θεωρεί ότι το Green Deal είναι μια ευκαιρία είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταβούμε σε ένα οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Και νομίζω ότι ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολλά κρατημέλη που θα συμφωνήσουν μαζί μας. Να σχολιάσω επίσης ε, τις, αυτά τα οποία είπατε σχετικά με τις θέσεις της κρατικής κυβέρνησης για τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο ανεπίσημο υπουργικό που θα γίνει στην Κροατία. Η κυρία Ζαλέσκα έθεσε το ερώτημα. Και η κυρία Γιώργο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανεπίσημης συνάντησης ε, το βασικό θέμα θα είναι η βιοπικιλότητα. Η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα, η χρηματοδότηση της κλιματολογικής ή κλιματικής ουδετερότητας ε, και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα τρία θέματα για την ανεπίσημη συνάντηση. Για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, Έγινε παραπομπή, ε, αναφερθήκατε στα 16 ανθρακορχεία. Νομίζω ότι αυτό το ανέφεραν πάρα πολύ στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Και ε, ετέθηκε το ερώτημα ε, πώς μπορούν να συμβαστούν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι τα άτυπα Υπουργικά Συμβούλια είναι το ιδανικός φορέας έτσι ώστε να γίνει συζήτηση για την κλιματική ευδετερότητα, για το μέλλον της Ευρώπης και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή, να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις συζητήσεις το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα βεβαίως ε, πολλά κράτη δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ε, ε, θετικά κίνητρα στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά το βασικότερο είναι να τα συμπεριλάβουμε, να μην τα αποκλείσουμε. Το να τα αποκλεί κανείς από την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό δεν είναι σωστό. Και εσείς το είπατε, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα, ότι αυτά τα 16 ανθρακοριχεία προκαλούν τόσο μεγάλη ρήπανση όσο τα 250 ανθρακοριχεία στο υπόλοιπο της Ευρώπης, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όσον αφορά την συμφωνία για τα Καρπάτια, ετέθηκε αυτό το ερώτημα. Ε, πράγματι, εμείς κατανοούμε ότι πρέπει να προστατευτεί αυτή η περιοχή και θέλουμε να ε, δείξουμε ενδιαφέρον συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και κατόπιν ετέθηκε ένα θέμα σχετικά με τις ε, ορμόνες ενδοκρινικοί διαταράκτες και ε, θα αποφασίσουμε ε, πώς θα προχωρήσουμε. Αυτά θα τα αποφασίσουμε μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Κρίστεν έθιξε ένα θέμα ε, σχετικά με την κυκλική οικονομία. Ε, προτάθηκε ένα νέο πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία. Ε, βεβαίως όλοι μας γνωρίζουμε και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει με αυτό το πρόγραμμα δράσης να διασφαλίσει να περάσουμε πράγματι σε μια κυκλική οικονομία. αυτή, αυτός ο όρος, κυκλική οικονομία, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, ε, συζητιέται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε μονομένα κράτη-μέλη. η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η κυκλική οικονομία, αυτά τα δύο θέματα αλληλοσυμπληρώνονται και ε, αυτούς τους στόχους ίσως μπορούμε να τους επιτύχουμε μέχρι το 2050. Αυτά τα θέματα τα προβλέπουμε για το ε, Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Ιουνίου και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η κατάλληλη χρονική στιγμή. το θέμα των σχέσεων ε, μεταξύ ε, της ΚΟΠ που θα λάβει η χώρα στην Κίνα. Πράγματι το θίξατε αυτό και πράγματι ε, υπάρχει έντονη προετοιμασία για μία σειρά πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμφωνώ απόλυτα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις τώρα παρουσιάστηκε η Πράσινη Συμφωνία, αλλά θα πρέπει να δημοσιευτούν και πολλές ε, άλλες ε, συμφωνίες. Ε, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δεσμευτούμε και θα εργαστούμε σκληρά για την προετοιμασία της ΚΟΠ στην Κίνα και αυτές τις ε, συζητήσεις ε, θα τις ε, έχουμε κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης στο Split. Γιατί με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε μέχρι τον Ιούλιο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Κατόπιν, η κυρία Γκλάμπακ έθιξε το θέμα της στρατηγικής. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια νέα στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και εμείς ε, θα προσχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση ακριβώς όπως θα συμβεί και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. τέθησαν ε, διάφορα θέματα για την ε, βιοπικιλότητα, ότι ε, θα πρέπει να διδεθούν περισσότερα κονδύλια για την βιοπικιλότητα. Το έχω ήδη πει, δυστυχώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Υπουργών Περιβάλλοντος, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε στις ε, επίσημες και ανεπίσημες συζητήσεις μας και αυτή την ευαισθητοποίηση μπορούμε να την μεταφέρουμε και σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να είναι γνωστό ε, πόσο επίγοντα είναι τα μέτρα για την ε, βιοπικιλότητα και τη χρηματοδότησή της. Έχουμε λοιπόν την Πράσινη Συμφωνία και ένα κομμάτι αυτής αφορά την ε, χρηματοδότηση της ε, βιοπικιλότητας. Ε, και το επόμενο ερώτημα που ετέθη από τον Κροάτη συνάδελφο δεν εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες και γι' αυτό δεν θα εξεταστεί από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε αυτά μεταξύ μας σε άλλου τύπου συναντήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Θα συνεχίσουμε στις 2.30.